του Προέδρου. Η σημερινή συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά μέσω ίντερνετ, web streaming. Υπάρχει διαθέσιμη διερμηνία σε 16 γλώσσες. Και τώρα θα ήθελα μισό λεπτό την προσοχή σας, γιατί υπάρχει μια τροποποίηση του ε, κανονισμού για την κοινή ΚΟΑ 1308-2013. Ε, η Γενική Διεύθυνση της Προεδρίας, το αντίστοιχο τμήμα για τις αλλαγές του κανονισμού, μας ενημέρωσε ότι υπάρχει διορθωτικό έγγραφο για τον ε, κανονισμό για την ε, ΚΟΑ 1308 του 2013 μετά από τη διαπίστωση ότι υπήρχε ένα τεχνικό σφάλμα. Ε, σας έχει διαβιβαστεί αυτό με τα έγγραφα της συνεδρίασης, το Κοριγέντου και στο άρθρο 141, παράγραφος 2, ο όρος ισογλυκόζη είχε προσθεθεί κατά λάθο κατά την ε, τελική οριστικοποίηση του κειμένου. Θα πρέπει να διαγραφεί ο όρος αυτός, διότι δημιουργεί ε, περιττές υποχρεώσεις για τους ε, ενδιαφερόμενους του τομέα. Αλλά επειδή η διόρθωση αυτή αφορά όλες τις γλωσσικές εκδοχές, η τροποποίηση πρέπει να εγκριθεί επισήμως στην Ολομέλεια. Εάν η Επιτροπή μας συμφωνεί για την τροποποίηση, η έγκριση θα γίνει στη διάρκεια της επόμενης ε, ολομέλειας του Στρασβούργου. Συμφωνείτε, υπάρχουν παρατηρήσεις, όχι, πολύ καλά. Συνεχίζουμε. Δεύτερη σημαντική ανακοίνωση, θα ήθελα σας παρακαλώ να σας ζητήσω όλους να έρθετε σε ένα αποχαιρετιστήριο κοκτέιλ που θα κάνουμε εδώ έξω από την αίθουσα για να γιορτάσουμε μαζί το πέρας ε, μιας ε, σημαντικής θητείας. Όλοι οι συνάδελφοι της Επιτροπής ε, Γεωργίας, εδώ απ' έξω λοιπόν στις 6.30. Τρίτη ανακοίνωση. Έκθεση Πυρίλο. Για το κόστος των ελέγχων. Θα θυμάστε όλοι ότι η Επιτροπή μας είχε υπερψηφίσει μία τροπολογία προκειμένου να εξαιρεθεί η γεωργία στις ε, δαπάνες ε, για τους ελέγχους. Αυτή η τροπολογία, την οποία υπερψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία η Επιτροπή μας, απορρίφθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Επομένως, ε, προετοιμαζόμαστε, κάνουμε συλλογή υπογραφών για να ε, ξαναπροτείνουμε την τροπολογία στην Ολομέλεια. Δεν ε, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Χρειαζόμαστε όμως 40 τουλάχιστον υπογραφές. Δεν υπάρχει δυνατότητα να υποβληθεί ως Επιτροπή γιατί έχει εκπνεύσει προθεσμία γι' αυτό. Θα ήθελα όμως να σας ζητήσω να υποστηρίξετε αυτή την τροπολογία και να υπογράψετε γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξαιρεθεί η γεωργία. Γνωρίζετε άλλωστε ότι οι γεωργοί ε, έχουν ε, ε, πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ερεσιμότητα Ο κύριος Ντες. Ο κύριος Δες. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, αγαπητέ Κάρλο. Ακριβώς επί του σημείου αυτού επειδή θα πρέπει να υποβληθεί στην Ολομέλεια, υποστηρίζω απολύτως αυτή την πρότασή σου και στην ομάδα μου θα προσπαθήσω να λάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες υπογραφές. Ας είναι και περισσότερες από 40, τόσο το καλύτερο. Θα έκανα λοιπόν μια έκκληση και στις άλλες ομάδες να συνυπογράψουν όσο το δυνατόν περισσότεροι ώστε να μπορέσουμε να το υποβάλουμε στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ, Άλμπερτ. Δεν έχει έρθει ακόμα ο Λουί Καπούλα Σάντο. Το συζητήσαμε στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Αν κατάλαβα, θα υποστηρίξουν η Μπρίτα. Να δούμε, να δούμε τι θέση θα λάβουν οι συνάδελφοί μου. Πιστεύω ότι αρκετοί θα το υποστηρίξουν αυτό και θα παρεκκλίνουν τις προηγούμενες γραμμές τους. Αρκετοί. Ευχαριστούμε, Μπρίτα. Χωρίς Πρόεδρος. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Προχωρούμε λοιπόν. Ε, σημείο 3. Ανταλλαγή απόψεων για την κρίση της Αφρικανικής Πανόλης των Χείρων και το ρωσικό εμπάργο στο χείριο κρέας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινά λοιπόν η σημερινή συνεδρίαση με μια συζήτηση για τον ευρωπαϊκό ε, τομέα χείριου κρέατος η συζήτηση αυτή έχει προκύψει από τα αρκετά περιστατικά αφρικανικής ε, πανόλης των χείρων σε χείρους από τη Λιθουανία και την Πολωνία. Παρά το γεγονός ότι είναι περιορισμένα τα περιστατικά και ε, λήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού της, ε, του φαινομένου βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η Ρωσία έχει επιβάλει απαγόρευση όλων των εισαγωγών ε, χείριου κρέατος από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό φυσικά δημιουργεί σημαντικές αναταραχές ε, στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εδώ ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Λάντισλαβ Μίκο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, ο οποίο θα απαντήσει στις ερωτήσει μα για την παρούσα κατάσταση και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο, στον κύριο Σεκεριέσκη, ο οποίο ε, μα ζήτησε να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση για το θέμα αυτό. Παρακαλώ κύριε Σεκεριέσκη, έχετε το λόγο και στη συνέχεια θα ακούσουμε του υπολείπου και μετά θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μίκο για να απαντήσει στι ερωτήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα από την αρχή να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα αυτή να γίνει η συζήτηση στην Επιτροπή μας στο, για του σημαντικού αυτού θέματος. Όπως είπατε και εσείς τα τέλη του Ιανουαρίου επειδή υπήρξαν δύο κρούσματα αφρικανικού πυρετού των χείρων στη Λιθουανία, η Ρωσική Ομοσπονδία απαγόρευσε τις εξαγωγές μας χειρίου κρέατος είχαμε <clears throat> από το σύνολο της Ένωσης, απαγόρευση της εισαγωγές. Επίσης, δύο κρούσματα εμφανίστηκαν στην Πολωνία με αγριοχούρουνα. Η ρωσική απαγόρευση λοιπόν εφαρμόστηκε παρά το γεγονός ότι η Πολωνία και η Λιθουανία μέσω έλαβαν μέτρα αντιμετώπισης της διάδοσης του ιού σύμφωνα με τους κανόνες της Διεθνούς Οργάνωσης ε, Υγείας δεν ευθύστηκαν νέα κρούσματα και είναι γνωστό ότι ο Αφρικανικός πυρετός των χείρων δεν θέτει κίνδυνο ε, ε, για τους ανθρώπους. Άλλες χώρες μέλη άρχισαν να συζητούν μονομερός με την Μόσχα πράγμα το οποίο σημαίνει ότι παραβιάζουν τις αρχές της ενωσιακής αλληλεγγύης και των κανόνων του ενιαίας αγοράς. Να ε, μην ξεχνάμε ότι οι με τέτοιο σκληρό διαπραγματευτή όπως η Ρωσία απαιτούν μια ενιαία στάση εκ μέρους της Ένωσης. Το ρωσικό εμπάργκο που άρχισε να εφαρμόζεται πριν από δύο μήνες δεν έχει καθόλου μειωθεί, ούτε βλέπουμε προοπτικές συμφωνίας η παραγωγή και εξαγωγή χειρίου κρέατος από την Ένωση Εν τω μεταξύ υπέστησαν ζημίες εκατομμυρίων ευρώ κάθε εβδομάδα, εφίστανται. Κάθε πρόσθετη μέρα εφαρμογής του εμπάργου σημαίνει ότι θα εμβαθύνεται η κρίση. Μερικοί έμποροι και παραγωγοί είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και αρχίζουν τις απολύσεις. Λόγω του εμπάργου ακριβώς. Επίσης έχει πέσει πολύ η τιμή του χειρίου κρέατος και στις 2 Απριλίου, την περασμένη εβδομάδα δηλαδή, η Ομοσπονδιακή, το, ε, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εποπτείας της Ρωσίας μας πληροφόρησε ότι από σήμερα 7 Απριλίου θα αρχίσει η Ρωσία να, επεκτείνει, να παρατείνει το εμπάργο, να το επεκτείνει όχι μόνο προς την Πολωνία και Λιθουανία και ούτε μόνο για ζώντες χείρους αλλά και για μεταποιημένο χείριο κρέας. Αυτό σημαίνει, ε, σας επαναλαμβάνω ότι αρχίζει από σήμερα να εφαρμόζεται η απόφαση αυτή και για τα μεταποιημένα χείρια προϊόντα που δεν θα μπορούν να εξάγονται από την Πολωνία και τη Λιθουανία προς την Αρασία. Θα ήθελα να ακούσω τις εξηγήσεις περί αυτού της Κομισιόν και να τη συζητήσω να λάβει μέτρα ώστε τέτοια άνηση μεταχείριση να παρεμποδιστεί. ειδικά για την Πολωνία και τη Λιθουανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρίε και κυρίε και να ξεκινήσει η συζήτηση. Τρει συνάδελφοι προ το παρόν έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριο ε, Βατσεπόσκοφσκι, ο κύριο Γέρ, ο κύριο Βατσεκόφσκι καταρχά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι, είναι αλήθεια ότι από σήμερα ισχύει μια ολική καθολική απογόρευση εισαγωγής χείριου κρέατος στη Ρωσία από την Πολωνία. Αυτό μας ανακοίνωσαν οι αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και αναρωτιόμαστε εάν τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοινή αγορά ή όχι. Διότι εάν η Ρώσικη Ομοσπονδία μπορεί να διχάσει και να διαιρέσει την, την αγορά μας και να επιλέξει από πού και από ποιους θα παίρνει χείριο κρέας ή όχι, αυτό σημαίνει ότι τελικά δεν έχουμε μία ενιαία αγορά στην Ευρώπη, αλλά ένα συνοθήλευμα 28 διαφορετικών αγορών. Γι' αυτό ζητούμε εντόνως από την Εκτελεστική Επιτροπή να δράσει ταχύτατα για να μην επιτρέψουμε την περαιτέρω διάσπαση στα εξών συνετές δηλαδή η ευρωπαϊκή ε, κοινή αγορά. Και αυτό θίγει ιδιαίτερα και ε, μερικές καινούργιες ε, χώρες που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ε, την κατάσταση αυτή για να κερδίσουν χρήματα ε, προς ίδιο όφελος και αυτό πρέπει να το τονίσει πολύ αυστηρά η Κομισιόν διότι εδώ διακυβεύεται η αρχή της αλληλεγγύης. Αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι αυτή την αφρικανική πανόλη των χείρων η οποία μην ξεχνάμε για πρώτη φορά διαπιστώθηκε στη Ρωσία και διαδίδεται, μεταδίδεται από τη Ρωσία προς τα έξω. Όχι αντίθετα, προς την αντίθετη κατεύθυνση, από τη Ρωσία προς τα έξω, προς άλλες χώρες. Στην Πολωνία υπήρχαν δύο περιπτώσεις ε, ε, που επισημάνθηκαν ε, σε αγριόχειρους, όχι σε εκτροφία χείρων πιστεύουμε λοιπόν ότι η Ρωσία προσπαθεί να τιμωρήσει την Πολωνία για τη στάση που κράτησε κατά την κρίση της Κρυμαίας. Αυτά έχω να πω από τη δική μου πλευρά. Αυτή είναι η άποψή μου και τώρα ειδού οι ερωτήσεις μου. Η Κομισιόν προβλέπει κάποια αποζημίωση προς τους παραγωγούς εκείνους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις προστατευόμενες ζώνες. Υπάρχουν παραγωγοί σε προστατευόμενες ζώνες, αλλά υπάρχουν και μερικοί και άλλοι εκτός, οι οποίοι πραγματικά ζημιώνονται πολύ λόγω της πτώσης, της μείωσης των τιμών του χοιρινού κρέατος. Ε, η πολωνική κυβέρνηση θα ήθελα να ξέρω, ζήτησε αποζημίωση, έκανε αίτηση αποζημίωσης προς την Κομισιόν και η Κομισιόν θα δεχτεί ή όχι μια, ένα τέτοιο αίτημα της Πολωνίας αν έγινε. Υπήρξε λοιπόν αίτημα αποζημίωσης από τους παραγωγούς που ζημιώθηκαν λόγω πτώσης των τιμών και η Κομισιόν θα το δεχόταν αυτό το αίτημα ή όχι. Ο Πρόεδρος. Η, η κυρία Γίγκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις για την ε, ε, την ιατρική υγιεινή την, και τα θέματα, τα παρεμφερή, τα οποία θα συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα στο Στρασβούργο, την ιατρικά θέματα θα πρέπει να σεβόμεσα τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα και, και ήθελα και εγώ να ρωτήσω την Κομισιόν αν θα υπάρξει οικονομική ενίσχυση προς τους θυγόμενους εντός ή εκτός προστατευόμενων ζωνών είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να πλήξει οποιονδήποτε παραγωγό ή περιφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη. Υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι οι οποίοι με μία τροπολογία δεν δέχονται ε, μια τέτοια στρατηγική διότι πιστεύουν ότι σε περίπτωση μιας τετοια ζημιάς θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ένα κράτος μέλος να υπεραμεινθεί των συμφερόντων του και να δράσει μεμονωμένα. Ε, αυτό πιστεύουν ε, ότι επαφίεται στη διεκριτική ευχέρεια των κρατών ε, μελών και ότι αν ένα κράτος είναι αρκετά δυνατό μπορεί να δράσει από μόνο του. Ε, γι' αυτό σας παρακαλώ θερμά να μην υπερψηφίσετε αυτή την τροπολογία για μεμονωμένη δράση, αλλά να δείξετε όλη την απαραίτητη αλληλεγγύη. Η, η Μπρίτα και μετά ο Καλινόφσκι. Η Μπρίτα. Ευχαριστώ αυτό το, το θέμα, το καυτό θέμα της εμπορικής πολιτικής και της Ρωσίας γίνεται όλο και συχνότερο ε, με την πανόλη των χείρων, με προηγούμενες ε, με προηγούμενα προβλήματα ε, ε, εκτροφής ζώων. Ε, με το παραμικρό η Ρωσία κλείνει τα σύνορά της, απαγορεύει τις εισαγωγές κλπ. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπεται αυτό. Πρέπει να διαχωρίσουμε την φυτο και κτηνιατρική πολιτική από την εμπορική πολιτική υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικά, δύο διαφορετικές διευθύνσεις στην Κομισιόν και ρωτώ την Κομισιόν μπορούν τώρα αυτές οι δύο εντελώς ξεχωριστές διευθύνσεις να συνεργαστούν ιδιαίτερα στο θέμα της Ρωσίας που έχει προκύψει τώρα. Ευχαριστώ Καλινόφ και μετά ο κύριος Ντές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν από μια εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες ε, και οι υπηρεσίες ε, φυτοϊγείας από τη Ρωσία προσέγγισαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ζήτησαν να διαβιβάσει ένα κατάλογο φυτών από διάφορα κράτη-μέλη και να μην, ε, που αγοράζουν ζωοτροφές για ε, την Πολωνία για να χρησιμοποιούνται ε, για κατανάλωση χειρινών. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι σκοπεύετε να κάνετε. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ξεκινήσει μια διαδικασία ε, στον ΠΟΕ για το θέμα αυτό, αλλά τι γίνεται με τους Ρώσους. Εάν τηρήσουν από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτά τα οποία ζητάει η Ρωσία, αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία έχει επιτύχει τον πολιτικό της στόχο και φυσικά θα δημιουργήσει ε, αναταραχή μεταξύ των κρατών μελών. Ουσιαστικά παρεμβαίνει στα πολιτικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, ε, αυτό ακούστηκε και αλλού σήμερα, Ο κώδικας του ΠΟΕΗ λέει ότι η περίοδος επόασης της συγκεκριμένη νόσου είναι 15 ημέρες. Εάν δεν υπάρξουν λοιπόν νέα περιστατικά στην Πολωνία και στη Λιθουανία, σημαίνει ότι ο ιός δεν έχει ε, μεταδοθεί σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ρωσία μέχρι τούδε τήρησε τα ε, πρότυπα και δεχόταν όλες αυτές τις ε, οδηγίες του ΠΟΗ ε, και επέτρεπε επεξεργασμένο μεταποιημένο κρέας να εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εξαίρεση τις συγκεκριμένε ε, περιοχές. Η ερώτησή μου είναι τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αίτημα που έθεσε η Ρωσία και τα θέματα τα οποία ε, ρώτησαν και οι συνάδελφοι για τις αποζημιώσεις και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Καλινόφσκη, ο Άλμπερτ Ντες και μετά ο κύριος Όριτσικ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρέπει να προσέξουμε σε αυτό το θέμα να παραμείνουμε αλληλέγγυοι στην Ευρώπη. Ξέρω ότι από τον τομέα του γάλακτος οι κυρώσεις είναι αυθαίρετες. Η Γερμανία είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος με 16 κρατήδια και ο συνάδελφος κύριος Σικέρσκι ξέρει πολύ καλά ότι ορισμένα ομοσπονδιακά κρατήδια ε, είχα, υπήρξαν σήματα μιας απαγόρευσης εξαγωγών, ε, εισαγωγών αν θέλετε, αλλά όχι. Λοιπόν, με αυτό το ομοσπονδιακό σύστημα βλέπετε ότι μπορούν να γίνουν πολλές αυθαιρεσίες στην εμπορική πολιτική. Και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το αποφύγουμε. Έχω και μια άλλη ερώτηση για την Κομισιόν. Πώς θα, τι θα γίνει με την περαιτέρω εξέλιξη τη κατάστασης στην Ουκρανία. Η Ρωσία θα λάβει, εάν λάβει νέα μέτρα, υπάρχει μεγάλος ε, κίνδυνος του μποϊκοτάζ από πλευρά δύση προς τη Ρωσία. Οπότε, ε, πώς θα ζητήσουμε εμείς στη, στη, στη Ρωσία να αλλάξει στρατηγική όταν εμείς θα ε, επιβάλλουμε πολύ αυστηρά ε, εμπάργο με πολύ μεγάλες επιπτώσεις ενδεχομένως στην περίπτωση της Ουκρανίας. Θα με ενδιαφέρε λοιπόν μια τέτοια... Ε, πώς θα είναι η προσέγγιση αυτή της, της ενδεχόμενης κατάστασης στο μέλλον, εάν εμείς μποϊκοτάρουμε τελικά και απαγορεύσουμε και, και επιβάλλουμε μποϊκοτάζ έναντι της Ρωσίας. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου είναι αντίστοιχη και αφορά τα θέματα της ελληνικής. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχει στοιχεία για τις εξαγωγές προς τη Ρωσία χείριου κρέατους και μεταποιημένου χείριου κρέατος. Υπάρχουν άλλες χώρες πέραν της Πολωνίας και της Λιθουανίας ε, στις οποίες να επιτρέπεται ακόμα η εξαγωγή προς τη Ρωσία ή το εμπάργο της Ρωσίας αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τι συμβαίνει εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αναφέρομαι στην περίπτωση του ε, αποθηκευμένου κρέατος στη Ρωσία αν μειώνονται τα ποσοστά των ε, ε, αποθεμάτων ε, χείρου κρέατος, τι ακριβώς κάνει η Ρωσία για να το τα στοιχεία της. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ. Ξέρουμε ότι η Ρωσία σε τέτοιες ε, περιπτώσεις που ε, υπησέρχονται θέματα ακτινιατρικά, προστασία της υγείας, δημόσιας υγείας, ασθενειών, των ζώων κλπ. Και βεβαίως αυτά άπτονται άμεσα των εμπορικών ε, συμφωνιών και συναλλαγών. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Κομισιόν πώς πάνε οι διαβουλεύσεις με τη Ρωσία, τι γνωρίζει περαιτέρω η Κομισιόν, γνωρίζει ότι κινούνται ορισμένες στα παρασκήνια ορισμένα κράτη-μέλη με δική τους πρωτοβολία ε, για να ε, διορθώσουν την κατάσταση και τι σκέφτεται να πράξει η Κομισιόν επ' αυτού. Ε, έχει ενδείξει η Κομισιόν ότι ορισμένα κράτη-μέλη προσπαθούν να περάσουν τη δική τους στάση, τη δική τους βούληση. Έχει απευθυνθεί σε αυτά τα κράτη η Κομισιόν, έχει κάνει κάποια παρατήρηση, κάποιο διάλογο διότι ε, εν συνεχεία πηγαίνουμε σε άλλα χωράφια προς την εξωτερική πολιτική και παρεκκλίνουμε. Δηλαδή μέσω της εσωτερικής αγοράς και της τρευλώσεων που ενδεχομένως συμβαίνουν ε, φτάνουμε και στην εξωτερική πολιτική. Πρέπει να έχουμε εμείς μια στρατηγική η οποία είναι διαφανής, συνεκτική και ε, αλληλέγγυη. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε Πέτερ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μίκο για να απαντήσει στις ερωτήσεις, να μας δώσει και κάποια νεότερα σχετικά με το εμπάργο από πλευρά Ρωσίας. Παρακαλώ, Μίκο. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα προσπαθήσω More light on... Uh, να σας απαντήσω όσο μπορώ καλύτερα. Καταρχήν, η Κομισιόν είχε στενές επαφές με τη ρωσική πλευρά από την αρχή και ακόμα και νωρίτερα γιατί ο Αφρικανικός πυρετός των χείρων άρχισε στη Γεωργία πριν από πολλά χρόνια και έφτασε μέχρι το βάθος της Ρωσικής Ομοσπονδίας πριν να φτάσει στα σύνορα της Ένωσης και είχαμε επιμείνει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα το έδαφος της Μπελαρούς και της Ρωσικής Ομοσπονδίας προσφέραμε μάλιστα και χρηματική βοήθεια για την εφαρμογή αυτών των μέτυρων. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι οι συνομιλητές μας από τη Ρωσία δεν κατάφεραν να εμποδίσουν την επέκταση αυτή του χειρίου πυρετού και έχουμε στοιχεία ότι πάνω από χίλια κρούσματα υπήρξαν αφρικανικού χειρίου πυρετού πέρυσι στη Ρωσία και τη Λευκορωσία σε σύγκριση με τέσσερα κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιθουανία και Πολωνία με αγριοχείρους. Έχουμε λοιπόν επαφές και σε τεχνικό επίπεδο και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και σε άλλα. Δυστυχώς όμως η προσέγγιση της ρωσικής πλευράς δεν ήταν πολύ επικαδαμητική. Ξέρουμε ποια εξαγωγικά συμφέροντα υπάρχουν και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα. Η Ρωσία μπήκε στον ΠΟΕ και υποσχέθηκε να είναι αξιόπιστος εμπορικός εταίρος με εφαρμογή των διεθνών προτύπων. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι η αντίδρασή τους είναι δυσανάλογη με τα γεγονότα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολόγηση για αυτά τα μέτρα. Εξάλλου η Ρωσία δεν λέει ότι πρόκειται για ολική απαγόρευση αλλά για πρόβλημα με τα πιστοποιητικά εξαγωγών και γι' αυτό δεν δέχονται καμία εξαγωγή διότι δεν είναι σωστά τα πιστοποιητικά. Εμείς αντιδράσαμε άμεσα όπως κάνουμε πάντοτε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και μηχανισμούς και προτείναμε την αλλαγή των πιστοποιητικών που δεν δεχόταν η Ρωσία αλλά κάθε φορά μας ζητούσαν όλο και περισσότερες τεχνικές πληροφορίες κλπ. κλπ. Δώσαμε, χορηγήσαμε όλες τις πληροφορίες που σχετικές και απαντάω εδώ στο ερώτημα του εάν όλα αυτά στρεβλώνουν τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό όταν υπάρχουν ευαίσθητες πληροφορίες ως προς τον ανταγωνισμό δεν τις δίνουμε στη ρωσική πλευρά. Τώρα γιατί υπάρχουν αυτά τα κρούσματα. Οι αγριόχειροι μάλλον διώχτηκαν, οθήθηκαν από την Λευκορωσία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του κυνηγιού που εφαρμόστηκε στη Λευκορωσία κατά των αγριοχείρων και γι' αυτό ξέφυγαν από τις περιοχές όπου ζούσαν σε άλλες πιο ήσυχες για αυτούς τους αγριόχειρους. Συζητήσαμε για αυτό το θέμα και με τους επιστήμονες αλλά δεν υπήρξε νέο κρούσμα και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η προσέγγιση μας που είναι η νομισμένη κάθε φορά ήταν η σωστή. Βέβαια η ρωσική πλευρά πάντοτε αρνείται να αναθεωρήσει την απαγόρευση των εμπάργων και καμιά φορά προτείνει και πρόσθετα μέτρα πολύ δύσκολα κατανοητά όπως ότι οι Ρώσοι θα σταματήσουν και τη μεταφορά χειρίου κρέατος από ολόκληρη την Πολωνία ενώ είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει τέτοια μεταφορά αφού δεν γίνονται οι εξαγωγές. Άρα δεν καταλαβαίνουμε καν τι σημαίνουν αυτές οι ανακοινώσεις από τη ρωσική πλευρά. Μάλλον είναι πολιτικά μέτρα και όχι τεχνικά και δεν έχουν καμία σχέση με την κατάσταση. Εξαντλήσαμε όλες τις πολιτικές και διπλωματικές οδούς και αποφασίσαμε να δράσουμε νομικά στα πλαίσια του μηχανισμού επιλύσεως διαφορών του ΠΟΕ και αρχίσαμε ζητώντας διαβούλευση καταρχήν. Σήμερα το ζητήσαμε από τους Ρώσους και η απάντηση θα δοθεί αύριο. Βεβαίως θελήσαμε να δούμε και ποιες είναι οι επιπτώσεις στην αγορά και για να καθησυχάσουν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί και έμποροι πρέπει να τους πούμε ότι τα συμφέροντά τους θα τα προασπίσουμε. Εδώ τέθηκε και το ερώτημα αν κάνουμε κάτι ως αποζημίωση για τους παραγωγούς. Πρώτον, η χρηματοδότηση που εγκρίναμε πέρυσι 2,5 εκατομμύρια ευρώ για συγχρηματοδότηση Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία και Πολωνία φέτος ένα εκατομμύριο παραπάνω για την, τον καθαρισμό και την αποτοξίνωση των εγκαταστάσεων και για να αποφευχθεί η σφαγή χείρων που είναι υποπτή για μόλυνση. Έχουμε συζητήσει και το θέμα της αποζημίωσης και συζητήσαμε με τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Γεώργ που ήδη χορήγησε βοήθεια στην Πολωνία για τις σφαγές χείρων 35 ευρώ ανά 100 κιλά κρέατος με ανώτατο όριο 20.000 τόνους. Αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν και αναδρομικά από την αρχή που εφαρμόστηκε τη εφαρμογής του εμπάργκο από τις 26 Φεβρουαρίου για χείρους που έχουν τραφεί, ανατραφεί σε μολυσμένες περιοχές. μπορούμε να περιμένουμε ότι τέτοιες αποζημιώσεις ανάλογες θα χορηγηθούν και για τη Λιθουανία. Τώρα για τις συνεννοήσεις μεταξύ χωρών μελών και την αλληλεγγύη. Πρέπει να σας καθησυχάσω. Η Κομισιόν γνωρίζει πολύ καλά ότι οι διμερείς επαφές με τη Ρωσική Ομοσπονδία δεν είναι η σωστή μέθοδος και πληροφορούμε τις χώρες μέλη πρώτον για την πρόοδο των συζητήσεων που κάνουμε ως Ένωση και στον ΠΟΕ με τη Ρωσία, αλλά επίσης επιμένουμε να μην γίνονται διμερείς συζητήσεις. Από την εμπειρία μας ξέρουμε ότι ακόμη κι αν είναι πειρασμός για ορισμένα κράτη-μέλη να συζητήσουν θυμερός υπονομεύει αυτό την γενική προσέγγιση της Ένωσης και δεν θα καταλήξει σε καμία λύση. Την περασμένη εβδομάδα πήγα στην έκθεση Αγκρομπάλτ στο Κάουνας στη Λιθουανία και με ρώτησαν εκεί Λιθουανοί και Πολωνοί για τις διμερείς επαφές που έλεγαν ότι του συζήτησαν οι Ρώσοι, ότι δηλαδή το πρόβλημα θα λυθεί με διμερή συμβόλαια. Αλλά δεν ισχύει καθόλου αυτό, είναι τελείως παράλογο. Νομίζω λοιπόν ότι πρόκειται για μια πολιτική προσπάθεια υπονόμευσης της ευρύτερης ενωσιακής προσέγγισης. Σας παρακαλώ λοιπόν όχι διμερείς δράσεις και αντιδράσεις αλλά ενωσιακές. Στο μηχανισμό επίλυση διαφορών του ΠΟΕ νομίζω θα δοθεί η λύση εν καιρό το δέοντι. Τώρα, τι θα γίνει αν η πολιτική κατάσταση εξελιχθεί περαιτέρω στην Ουκρανία μου είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω σε τι βαθμό συνδέονται αυτά τα θέματα. Θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι εργαλείο έχουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα των εμπορικών φραγμών. Και αν υπάρχει τίποτε νεότερο θα σας πληροφορήσω. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λάντισλαβ Μίκο της Γενικής Διεύθυνσης ε, ΣΑΝΚΟ. Νομίζω ότι ήταν πληρέστατες οι απαντήσεις του και να δώσω λοιπόν το λόγο στον Αντιπρόεδρο, στον κύριο Σικεδιέσκη. Α, κύριε και εσείς θέλετε το λόγο. Θα ήθελα να ρωτήσω μία ε, ερώτηση στη συνέχεια. Ρώτησε κάτι για την αποζημίωση των αγροτών εκτός από τις ε, περιοχές στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για άλλους ε, κτηνοτρόφους ε, οι οποίοι έχουν απώλειες λόγω μείωσης των τιμών. θα υπάρξουν κάποια μέτρα και υπήρχε και μία ερώτηση, μια, ένα ειδικό αίτημα της πολωνικής κυβέρνησης επί του θέματος αυτού. Σας ευχαριστώ το θέμα των αποζημιώσεων για ε, κτηνοτρόφους εκτός ε, της ε, περιοχής στις οποίες υπάρχουν τα κρούσματα δεν έχει ακόμα συζητηθεί. Είναι εξελίξει συζήτηση και κοιτάμε να δούμε σε ποιο βαθμό θα έχουμε απλώς την οικονομική στήριξη για τις πληγήσεις περιοχές. Δεν γνωρίζω τίποτα περί οποιασδήποτε απόφασης από τους συναδέλφους Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας. Το δεύτερο τμήμα του ερωτήματός σας ποιο ήταν? Ποιο ήταν Poland... Α, για την Πολωνία δεν ξέρω να σας πω. Δεν ξέρω αν έχει υποβληθεί επισήμω το αίτημα. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις εν εξελίξη. Ξέρω ότι το Υπουργείο ρώτησε τι δυνατότητες αποζημίωσης υπάρχουν. Γι' αυτό ακριβώ και είναι εν εξελίξη αυτές τις συζητήσεις. Ωραία, ευχαριστώ. Ο κύριος Εκυριέσκη για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την, τις απαντήσεις της. Νομίζω ότι έχουμε ορισμένες απόψεις, ορισμένα, καταλήξει ορισμένα συμπεράσματα για το μέλλον, αν αυτό το σενάριο επαναληφθεί ε, και εάν μας πήξει και πάλι έχουμε ορισμένα, καταλήξει ορισμένα συμπεράσματα σε υψηλό επίπεδο ότι πρέπει να κάνουμε. Ε, υπάρχουν λοιπόν διαδικασίες ε, τις οποίες ε, έχουμε λάβει υπόψη και για να υιοθετήσουμε σκληρότερα μέτρα αλλά και για να βοηθήσουμε τους παραγωγούς. Διότι κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε ένα δύσκολο σενάριο σαν και αυτό εδώ ποιος θα πληρώσει την ύφη τελικά ποιοι. Η παραγωγή μας. Αυτοί δεν είναι που πλήττονται. Αυτοί θα χάσουν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα, μια σαφή πολιτική η οποία θα βοηθήσει ε, τους παραγωγούς να μην ε, χάσουν το εισόδημά τους και τα απαραίτητα προς το ζήν. Διότι η τιμή του χείριου κρέατος έχει πέσει όχι μόνο στην Πολωνία και στη Λουθιουανία αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως σε διαφορετικό ποσοστό, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν πέσει οι τιμές και πρέπει να είμαστε έτοιμοι όταν συμβεί ένα τέτοιο σενάριο να το αντιμετωπίσουμε. Μια τέτοια περίπτωση. Τώρα, ε, βάσει της εμπειρίας που έχουμε, η πανόλη των χείρων μπορεί να εξαπλωθεί προς δυσμάς και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ο Πρόεδρος. Ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε λήξαν το συγκεκριμένο θέμα. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ και τον ε, Διευθυντή, τον κύριο Λάντι Θαυμίκο, για τις απαντήσεις που μας έδωσε. Και επειδή ε, πλησιάζουμε στις 5.30, πολύ γρήγορα να συζητήσουμε το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης ε, για την επίσκεψη της ε, αντιπροσωπείας μας στην ε, Βαυαρία στις 24 με 26 Μαρτίου με 28 Μαρτίου, συγγνώμη. Με χαρά λοιπόν θα ακούσουμε μια αναφορά για την επίσκεψή μας στη Βαβαρία. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον Άλμπερτ Ντες, ο οποίος διοργάνωσε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα επίσκεψη, η οποία έφερε στην επιφάνεια πολλά χαρακτηριστικά της ε, περιοχής, κυρίως όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος, του λυκίσκου και αρκετούς ενδιαφέροντες τομείς παραγωγής ε, βιοενεργειακών προϊόντων. Συμμετείχαν αρκετοί συνάδελφοι, οι οποίοι είναι και παρόντες, ο κύριος Τζιμ ε, Νίκολσον, ο κύριος Ντόρφαν, ο κύριος Άιλουαρτ, ε, ε, όλοι οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Γεωργίας αυτή την επίσκεψη και υπήρχαν και συναντήσεις με τον Βαβαρό Υπουργό, τον Χέλμουτ Μπρούνερ. Να δώσω το λόγο στον Αλμπερντές για να μας πει εντάχει ε, τι συνέβη στην επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στη Βαβαρία 26 με 28 Μαρτίου. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους να ετοιμάσετε τις καρτέλες σας γιατί αμέσως μετά θα περάσουμε στην ψηφοφορία στο σημείο 5 για τις ε, πληροφορίες για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων, την έκθεση της κυρίας Εράνς Καρσία. Παρακαλώ, Άλπερτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα ε, ότι αυτή η επίσκεψη ε, που είναι και η τελευταία αντιπροσωπείας μας ε, κατά την θητή αυτού του κοινοβουλίου έγινε στη Βαβαρία. Ευχαριστώ όλους τους επικεφαλείς, όλους τα μέλη της αντιπροσωπείας και τους διερμηνείς, όλους όσοι συμμετέσχουν. Κύριε Πρόεδρε, εδώ γίνεται πολύ βαβούρα. Φασαρία. Φασαρία. Γιατί. Παρακαλώ, κάντε ησυχία, λέει ο Πρόεδρος. Μάλιστα. Λοιπόν, επισκεφθήκαμε τη Βαβαρία που από απόψε εδαφική επικράτεια είναι το μεγαλύτερο κρατήδιο, πάνω από 3 εκατομμύρια εκτάρια. Ε, 8,2 εκατομμύρια εκτάρια είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, επίσης χορτολιβαδικές εκτάσεις φτάνουν μαζί σε περίπου 9,5 εκατομμύρια εκτάρια, καλλιεργούμενες εκτάσεις και χορτολιβαδικές. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς ε, λειτουργεί όλη η υποδομή της γεωργίας ε, με την ε, συνεργασία σε θέματα υποδομών αλλά και χρήσης μηχανημάτων και στο Μιλχάουζεν έχουμε μια εξαιρετικά μοντέρνα, σύγχρονη ε, καλλιέργεια λυκίσκου και μεταποίησης του λυκίσκου. Επίσης όσον αφορά την ε, κράμβη, 4 εκατομμύρια ένα εκτάριο. Ε, ε, και ε, προωθούνται αυτές οι καλλιέργειες του Λυκίσκου και της ε, Κράμβης ιδιαίτερα 200 τρακτέρ έχουν μεταποιηθεί με μία απλή τεχνολογία έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν και στις εκτάσεις που καλλιεργούν κράμπι και στις εκτάσεις που καλλιεργούν λυκίσκο. Έχουμε λοιπόν μία συνεργασία των παραγωγών και συνεταιρισμό των παραγωγών για την μεταποίηση και προσαρμογή και χρήση των μηχανημάτων η οποία έχει ε, αποβεί πάρα πολύ θετική όσον Φορά τα εισοδήματά τους, το, το όφελος. Επίσης στην παραγωγή πατάτας 47 παραγωγοί έχουν ενώσει τις προσπάθειές τους για τη μεταποίηση της ε, πατάτας ε, έχουμε επίσης επισκεφθεί, επισκεφθήκαμε μία φάρμα η οποία έχει 80 γαλακτοφόρες αγελάδες. Η οικογένεια αυτή έχει πέντε κόρες ε, οι οποίες όλες σπουδάζουν αλλά εν συνεχεία μετά τις σπουδές τους τα κορίτσια αυτά είναι πρόθυμα να εργαστούν και να χρησιμοποιήσουν χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία τους στην ε, παραγωγική μονάδα των γονιών τους. Επίσης, ο κύριος ε, Μάιερ από την εταιρεία Bayernland μας εξήγησε το συνεταιριστικό προφίλ ε, της γαλακτοπαραγωγής, διότι 50% της παραγωγής γάλακτος στη Βαυαρία προέρχεται από συνεταιριστικές μονάδες και περίπου 40% από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εν συνεχεία στο Ούμπερβαλ επισκεφθήκαμε ε, μία μονάδα από τρεις νέους παραγωγούς, 210 εκτάρια και παράγει βιοαέρια, τα οποία χρησιμοποιούνται ε, για την ε, χρησιμοποίηση της ενέργειας σε τεράστια θερμοκήπια παραγωγής αγκουριών. Επίσης, ε, όσον αφορά τη Βίνη, ε, ε, επισκεφθήκαμε και μονάδες καλλιέργειας Βίνης, παραγωγικές μονάδες, πάλι συνεταιριστικές, οι οποίες λαμβάνουν και ορισμένε επιδοτήσεις από το εθνικό επίπεδο, κρατικό δηλαδή. Επίσης, επεξεργάζονται νέους σπόρους, κάνουν μία έρευνα για τη χρησιμοποίηση νέων σπόρων για την παραγωγή πιο αποδοτικών φυτών. Πήγαμε βεβαίως και σε ένα ζυθοποιείο, διότι δεν μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τη βαβαρική μπύρα. Την Παρασκευή υπήρχε ένα, ήταν μια ημερίδα βαβαρικής ε, γεωργίας ε, και συναντηθήκαμε με πολλούς παραγωγούς, αγρότες και είχαμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ε, συναντήσαμε και τον Κέρχαρτ, ο οποίος ζει στο Μόναχο και χάρηκε ιδιαίτερα που ξανασυνάντησα την ομάδα μας. Αυτή ήταν λοιπόν μια σύντομη παρουσίαση των, ε, της επίσκεψής μας, του προγράμματός μας στη Βαβαρία και περάσαμε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Άλμπερτ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση. Ε, υπάρχει και μια αναφορά για την αποστολή μας στη Βαβαρία, για όποιον θέλει να τη διαβάσει, σας έχει διανεμηθεί. Και τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, μισό λεπτό προσοχή, συνάδελφοι. Θα συζητήσουμε το σημείο 5 ενέργειες ενημέρωσης σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και προώθησή του στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Άγνιου, όχι για αυτό το σημείο. Παρακαλώ. Κύριε Άγνιου. Πρόεδρε, με αυτή την ευκαιρία θέλω πρώτον να σας ευχαριστήσω για τα τελευταία πέντε χρόνια που, μας, που μου δίνατε χρόνο ομιλίας ενώ συνήθως διαφωνώ με τους υπόλοιπους. Θα ήθελα όμως να σας δείξω εδώ μία γεωργό που λέγεται Liz Buckle και θα παρατηρήσετε ότι έχει μεγάλη αναπηρία στα χέρια διότι η μητέρα της κατά την εγκυμοσύνη πήρε θαλιδομίδι για, κατά της ναυτίας αυτή είναι τυχερή βέβαια γιατί πολλά από τα θύματα της θαλιδομήνης δεν έχουν ούτε χέρια ούτε πόδια. Δεν έχει πληρωθεί βέβαια πολύ αποζημίωση αλλά όσο μεγαλώνουν τα θύματα της θαλιδομίδης χειροτερεύουν τα προβλήματά τους και χρειάζονται περισσότερη στήριξη, περισσότερα χρήματα. Οι κατασκευαστές της θαλιδομίδης είναι μια γερμανική εταιρεία που λέγεται Grunenfold που θεωρεί ότι έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. εγώ διαφωνώ και πιστεύω ότι η γερμανική κυβέρνηση και η εταιρεία Grunenfold πρέπει να πληρώσουν περισσότερα. 30 λεπτά το χρόνο για κάθε γερμανό φορολογούμενο θα έλυναν το πρόβλημα και το, αν ήταν 50 λεπτά το ποσό θα ε, λυνόταν το πρόβλημα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια αναφορά την οποία μπορείτε αν θέλετε να υπογράψετε και μετά το πέρας της συνεδρίασης έχουμε ένα κοκτέιλ απ' έξω όπου μπορείτε να υπογράψετε και να πάρετε και πληροφορίες. Ευχαριστούμε κύριε Άγνιου λαμβάνουμε υπόψη ε, την υπόδειξή σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, περνάμε στο σημείο 5. Ενέργειες ενημέρωσης σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και προώθησή τους στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες. Όπως ε, γνωρίζετε, έγιναν δύο τριμερείς διάλογες, ε, στους οποίους ε, η διαπραγματευτική μας ομάδα κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του θέματος. Πριν ε, από την ψηφοφορία στο κείμενο το οποίο συμφωνήθηκε, θα δώσω το λόγο στην κυρία Εράνς Καρσία για να μας παρουσιάσει τα σημαντικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας. Θα ήθελα όμως ταυτόχρονα, δίνοντάς της το λόγο, να υπενθυμίσω ότι θα υπάρξει μία ψηφοφορία και θα γίνει ηλεκτρονικά. Επειδή λοιπόν δεν έχουν ε, υποβληθεί όλοι οι αναπληρωτές στη γραμματεία, θα ήθελα να είστε λίγο προσεκτικοί στην ψηφοφορία, θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος προηγουμένου. Έστερ, έχει το λόγο όμω, πριν από την ψηφοφορία. Πε μα πω πήγε η διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι χαρά μου να μπορέσω να σας πω ότι μετά από τις ε, διαπραγματεύσεις ε, το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο καταλήξαμε σε συμφωνία καταρχήν την οποία υποβάλλουμε προς σήμερα. Τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία ε, είχαν απασχολήσει τους ευρωβουλευτές στην ψηφοφορία την προηγούμενη φορά μπόρεσαν να τα υποστηρίξουν οι τα μέλη της διαπραγματευτικής μας ομάδας και ε, στηρίξαμε και τα όσα ζήτησαν οι πολιτικές ομάδες. Οι πολιτικές ομάδες συμμετείχαν και στις, στις τριμερείς διαπραγματεύσεις και καμία από τις πολιτικές ομάδες ε, δεν ήταν αντίθετη για τη συμφωνία. Ε, κατά πάσα πιθανότητα ψηφίζοντας σήμερα θα μπορέσουμε πολύ γρήγορα να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κάποιος έχει ζητήσει ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα. Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε διανατάσεως χείρις, Χειρός, όχι ηλεκτρονικά. Συγγνώμη, διορθώνει και πάλι ο πρόεδρος, ηλεκτρονικά ένα, αλλά όχι μονομαστική κλίση. Όσοι είναι υπέρ της διαπραγμάτευσης, ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Μισό λεπτό γιατί πρέπει να επαληθεύσουμε. κιούς. Πέρα τη ψηφοφορία. Ωραία. Εγκρίνεται. Επομένως με πολύ μεγάλη πλειοψηφία κιόλα, μπορούμε να περάσουμε στην Ολομέλεια για να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Συγχαρητήρια στην κυρία Εράν Καρσία και σε όσους ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Okay. Okay. José Bové, oui, no, je... έχει ζητήσει το λόγο. Νομίζω ότι μετά από αυτή την ψηφοφορία για την ε, προώθηση προϊόντων εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό θα ήταν ε, η Επιτροπή Γεωργία του Κοινοβουλίου και ίσω και άλλοι ευρωβουλευτέ να συντάξουν συλλογικά μία επιστολή η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών για να τους πούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα προϊόντα με ονομασία προέλευσης και δεν δεχόμαστε τα όσα προτείνουν ε, σε επίπεδο διεθνών διαπραγματεύσεων για τα προϊόντα αυτά. Ε, μας διαβιβάστηκε το έγγραφο από τη γραμματεία της Επιτροπής μας και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ αυτών των προϊόντων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Ο κύριος Ντές έχει ζητήσει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ε, ε, μετά από αυτά που είπαν, που ελέγχθη, κοίταξε αγαπητέ συνάδελφε, ξέρω ότι έχει συμφωνήσει σε μια προηγούμενη απόφαση του Κοινοβουλίου του 2010. Τότε είχαμε αποφασίσει και πολύ λογικά, μετά από έτοιμά μας, ότι αγροτικές εισαγωγές επιτρέπονται μόνο εάν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά μας πρότυπα καταναλωτικά, κτηνιατρικά ε, και είχαμε τότε υιοθετήσει αυτή την απόφαση με πλειοψηφία. Έχουμε μία σαφή εντολή και είναι πολύ ισχυρότερη αυτή η απόφαση. Προς αυτήν πρέπει να παραπέμψουμε. Ισχυρότερη από μία επιστολή. Ευχαριστώ θα υπερψηφίσω, εγώ θέλω να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης κυρίας Γκαρσία. Είμαι υπέρ, αλλά δεν δούλεψε το μηχάνημά μου. Ωραία, ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Συνάδελφοι, να περάσουμε τώρα στο σημείο 6. Ε, κατοξουσιοδότηση κανονισμός Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού 1307-2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις του Γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο κοινή γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του εν λόγω κανονισμού. Συνάδελφοι, ψηφίζουμε λοιπόν την πρόταση να απορρίψουμε την πρόταση της Επιτροπής για την κατεξουσιοδότηση πράξη αυτή για τις άμεσες ενισχύσεις. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες οι οποίες αιτιολογούν την απόρριψη αυτής της πρότασης, οι οποίες επιβλήθηκαν και από τις πολιτικές ομάδες αλλά και από βουλευτές μεμονωμένα. Πριν περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους εσάς ότι βάσει του άρθρου 87α του κανονισμού, το ψήφισμα πρέπει να περιλαμβάνει και δέουσα αιτιολόγηση της ένστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως, προκειμένου να μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε το ψήφισμα, θα πρέπει να εγκριθεί τουλάχιστον μία αιτιολογική σκέψη. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν εγκριθεί καμία αιτιολογική σκέψη, το ψήφισμα καταπίπτει. Είναι σαφές σε όλους. Επομένως, θα ψηφίσουμε και εδώ ηλεκτρονικά. Allora, recital A. Ah, iniziamo Αιτιολογική σκέψη Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή, ε. Αιτιολογική σκέψη ε, Σ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη H. Υπέρ. H υπέρ ναι. κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Ι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη J υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη και υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη L. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη M. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη N. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη O. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη P. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Q, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη R, υπέρ, κατά, υπέρ για το R, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη S, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη T, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Q. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επειδή δεν υπάρχει αρκετή δεν υπάρχουν αρκετοί για να εγκρίνουμε το θέμα, δεν υπάρχει ψήφισμα, επομένως δεν θα υπάρξει ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τις κατά κατεξουσιοδότηση. Για τη συγκεκριμένη ε, πράξη κατεξουσιοδότηση. Περνάμε τώρα στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης εξουσιοδότηση κανονισμό τη Επιτροπή για τη συμπλήρωση του κανονισμού 1306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείριση και ελέγχου και του όρου απόρριψη ή ανάκτηση πληρωμών, καθώ και τι διοικητικέ κυρώσει που εφαρμόζονται στι άμεσε ενισχύσει, τη στήριξη τη αγροτική ανάπτυξη και την πολλαπλή συμμόρφωση. Ε, θα ψηφίσουμε όπω και στο προηγούμενο θέμα. Θα ψηφίσουμε διανατώσεως χειρός όλα όλες τις αιτιολογικές σκέψεις και αν δεν εγκριθεί καμία αιτιολογική σκέψη θα προχωρήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Υπέρ της αιτιολογικής σκέψης A. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη B. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη C. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη D. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη E. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη F. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη G. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη H. Υπέρ. υπέρ της AIDS, κατά, αποχές απορρίπτεται, αιτιολογική σκέψη I, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, αιτιολογική σκέψη J, υπέρ, κατά, έλεγχος, για την αιτιολογική σκέψη I. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη. Ε, συνεχίζουμε δυνατά στο χειρός. Το J, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη K, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και επομένως και σε αυτή την περίπτωση Καταπίπτει το ψήφισμα. Σημείο 8. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε καταξιοδότηση κανονισμών της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού 1306-2013 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ. Και εδώ διανατάσσεως χειρός ε, ξεκινούμε την ψηφοφορία για τις αιτιολογικές σκέψεις. Η γραμματεία μου λέει ότι θα μπορούσαμε να τις ψηφίσουμε unblock γιατί είναι όλα σε αιτιολογικές σκέψεις του κυρίου Άγνιου. Ψηφίζουμε unblock, συμφωνείτε? Ποιος είναι υπέρ? υπέρ. Για τις αιτιολογικές σκέψεις του κυρίου Άγνου. Εσείς θα έπρεπε κύριε Άγνου να υπερψηφίσετε. Κύριε Πρόεδρε. Καλύτερα να τις ψηφίσουμε μία-μία. Ε, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Μπ, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Σι. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δι. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ή. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προσπαθήσαμε να το ψηφίσουμε μπλοκ, δεν τα καταφέραμε, τέλος πάντων προχωρούμε. Σημείο 9. Κατά εξουσιοδότηση κανονισμών της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού 1306-2013 όσον αφορά τις δαπάνες για τη δημόσια παρέμβαση. Διανατάσσεως χειρός μία προς μία για να μην υπάρχει αμφιβολία. Α, αιτιολογική σκέψη α, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Β, υπέρ. Κατά, Αποχές απορρίπτεται. Σι Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. D. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ή. υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και εδώ λοιπόν δεν υπάρχει πλειοψηφία. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία ψηφοφορία. Σημείο 10. Κατεξουσιοδότηση κανονισμός για τη συμπλήρωση του κανονισμού 1305 για τη στήριξη αγροτική αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξη για τη θέσπανση μεταβατικών διατάξεων. Ψηφίζουμε και εδώ μία προς μία ο χειρός. Υπέρ τη αιτιολογική σκέψη A. Κατά. απόχέ απορρίπτεται. B. Υπέρ. Κατά. αποχέ απορρίπτεται. C. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται, D υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, E υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. F υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, G υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν έχουμε κάποια λογική σκέψη, η οποία έχει πλειοψηφία 11. Εδώ έχουμε καταξουσιοδότηση κανονισμό που αφορά τον τομέα των απορροκυπευτικών και των μεταποιημένων απορροκυπευτικών Και σε αυτή την περίπτωση ψηφίζουμε μία προς μία τις τροπολογίες A, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. B, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. C, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, D, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, E, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, F, κατά, αποχές απορρίπτεται, G, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. H υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεν υπάρχει πλειοψηφία. Προχωρούμε λοιπόν σημείο 12. εξουσιοδότης κανονισμός για τη χορήγηση ενίσχυσης για συνοδευτικά μέτρα στο πλαίσιο καθεστώτος προώθησης κατανάλωσης οπωροκεπιπτικών στα σχολεία. Διανατάσσεως χειρός μία προς μία. Υπέρ της A. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. B. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. E. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και εδώ δεν υπάρχει καμία πλειοψηφία. Σημείο 13. Κατά εξουσιοδότηση κανονισμός για τα προγράμματα στήριξης του τομέα ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. Μία, μία. Ε, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. Β, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Σ, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δι, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. ή υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Προχωρούμε. Σημείο 14. Δύο μέμειναν. Εδώ έχουμε ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα για τα οποία χορηγούνται ενισχύσει για την ιδιωτική αποθεματοποίηση. Ω συνήθως, ε, αιτιολογική σκέψη A υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. B υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. C υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. D υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται ή υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελευταία κατεξουσιοδότηση πράξη, σημείο 15 στην ημερήσια διάταξη για τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμποελοϊνικό τομέα. Και εδώ μία-μία, διανατάσεως χειρός, ξεκινούμε. Ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. B υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. C υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. D υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ή, υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν υπάρχει κάποια αιτιολογική σκέψη η οποία να έχει πλειοψηφία και με αυτό ολοκληρώθηκε όλο το θέμα της μεταρρύθμισης κοινή γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστούμε, συνάδελφοι. Ο κύριος Μπαβέ έχει ζητήσει το λόγο. Μετά από αυτή την, Μετά ψηφοφορία ή μάλλον την ε, κοροϊδία θα ήθελα να πω ότι δεν έχω ξαναδεί ποτέ τέτοιο πράγμα. Ενώ υπήρξε στον τριμερή διάλογο συμφωνία για την κοινή αγροτική πολιτική και για τις κατεξουσιοδότησης πράξης, μερικές ομάδες διαφώνησαν και διατήρησαν, επέμειναν στη θέση τους και έτσι ψήφισαν επίσης, όπως οι συντηρητικοί και για ορισμένες ψηφοφορίες και οι φιλελεύθεροι. Είναι όμως απαράδεκτη στάση του ΕΛΚ ο εκβιασμός που την τελευταία εβδομάδα προσπάθησε με την αμφισβήτηση των κατεξουσιοδότησης πράξεων που είχαν δεχτεί και οι ίδιοι προηγουμένως έπραξαν έναν εκβιασμό για να μειώσουν ακόμη περισσότερο την ΚΑΠ. Είναι απαράδεκτο και εκβιασμός κατά της Κομισιόν και λυπάμαι που ο Επίτροπος Τσόλος υποχώρησε σε, αυτό τον εκβιασμό. Όσοι επέμειναν στη θέση τους είχαν το δικαίωμα να το πράξουν, αλλά όσοι αντιτάχθηκαν στις ίδιες τους τις τροπολογίες νομίζω είχαν απαράδεκτη στάση. Ελπίζω να υπάρξει και κάποια απάντηση. Αυτή φυσικά είναι η προσωπική άποψη του κυρίου Μποβέ και τώρα να ακούσουμε την άποψη των υπολείπων συναδέλφων. Η κυρία Γέγκελ είχε ζητήσει το λόγο πρώτα, Γέγκελ και μετά ο κύριος Ντές. Ευχαριστώ πρόεδρο και τονίζω ότι εγώ καταψήφισα. Αγαπητέ συνάδελφε, αυτό το οποίο κάναμε και ζήτησα στο Στρασβούργο και συμφώνησε ο διαμεσολαβητής ήταν πρόταση βελτιώσεων των κειμένων, τα οποία δεν, ήταν, ε, είχα συμπεριληφθεί στις πολιτικές μας αποφάσεις. Επί τρεις εβδομάδες εργαζόμασταν με την Κομισιόν και η Κομισιόν είχε συμφωνήσει με τα αιτήματά μας. Θα κάνει μία δήλωση, σαφώς θα υπάρχει μία δήλωση η οποία θα δεσμεύει την Κομισιόν στην υλοποίηση αυτών τα οποία αποφασίσαμε και γι' αυτό θα πρέπει να υλοποιηθούν αυτά και από όλε τις περιφέρειες και να μην τροποποιήσουμε ξανά τίποτα. Σύμφωνα με το δικαίωμα, έχουμε το δικαίωμα αυτό βάσει τη συνθήκης τη Λισαβόνας και χρησιμεύσαμε ως παράδειγμα εμεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για εθνικούς, για τους εθνικούς μας βουλευτές, διότι οι εθνικοί μας βουλευτές τρώνε το ξύλο, όχι εμείς. Είχαμε λοιπόν επιτυχία στα σημεία αυτά τα οποία ζητήσαμε ε, και γι' αυτό εγώ καταψήφισα τον ίδιο μου τον εαυτό. Διότι εγώ πιστεύω αυτά τα οποία είχαμε αποφασίσει ήταν και τα σωστά. Ε, ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος. Γιάρ, Ιντές, Άγνιο και άλλοι. Ο, Πέ, ο Πέτερ, Πέτερ Γιάρ. Ευχαριστώ. Δεν καταλαβαίνω διόλο την παρέμβαση του κυρίου Μποβέ και τις επεξηγήσεις του. Έχουμε μία νομική πράξη την οποία πρέπει να σεβαστούμε και είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε αυτές τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Έχουμε και το δικαίωμα τις επαναπαραπέμψουμε. Έχουν λοιπόν ελεγχθεί αυτές οι πράξεις ε, δεν ε, ήταν ικανοποιημένοι, ε, έγινε διαβουλεύσεις με την Κομισιόν και εγώ πιστεύω ότι το αποτέλεσμα τώρα είναι θετικό διότι η Κομισιόν δεσμεύτηκε βάσει των αποφάσεων που είχαμε λάβει. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα διαχείρισης των κατεξουσιοδότηση πράξεων, πώς θα τις διευθετήσουμε στο μέλλον και πιστεύω ότι κάθε επίτροπος ε, καλά θα κάνει στο μέλλον να προετοιμάσει τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις αυτές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε ε, αν υπάρχει μια επαναπομπή τότε βεβαίως θα πρέπει να επανεξεταστεί και η πράξη. Τι λέει μέσα η κατεξουσιοδότηση πράξη. Εμείς το κάναμε αυτό, την εξετάσαμε. Τώρα, ε, συμφωνώ ότι μπορεί να μην συμφωνούν όλοι, αλλά μην ξεχνάτε ότι εμείς βασιστήκαμε στις προηγούμενες αποφάσεις. Ε, τώρα, αν κάποιος έχει επικρίσεις, ναι, το καταλαβαίνω, αυτό είναι ένα γνώρισμα της δημοκρατίας, αν υπάρχουν επικρίσεις ή σχόλια, αλλά εμείς παραμένουμε πιστοί στις θεμελιώδεις αρχές μας. Ο κύριος Ντες, λέει ο πρόεδρος. Ε, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ντέ, θα ήθελα να επενθυμίσω και στον κύριο Μποβέ και στου υπολείπου ότι προκάλεσαν τόσο πολύ συζήτηση αυτέ οι πράξει κατεξουσιοδότηση, ότι διότι κατά τη συζήτηση, τουλάχιστον κατά την άποψη των περισσότερων συναδέλφων, θεωρούμε ότι απομακρύνθηκαν από τη συμφωνία στην οποία είχαμε καταλήξει. Για παράδειγμα, στις πρωτεΐνες δεν είχαμε συμφωνήσει εμείς ε, για συντελεστή 0,3 που βρήκαμε στην πράξη κατά εξουσιοδότηση. Δεν αλλάζει λοιπόν η συμφωνία, ίσα ίσα είναι ο σεβασμός της πολιτικής συμφωνίας. Ο Άλμπερ Ντες και μετά ο κύριος Σάκνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε Μποβέ, δεν καταλαβαίνω διόλου την παρέμβασή σου. Οι πράσινοι πάντοτε επαναμείνονται της δημοκρατίας, της βασικής δημοκρατίας και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητεί τη δημοκρατική διαδικασία εδώ στο Κοινοβούλιο και δει από την ομάδα σου Έχουμε χρησιμοποιήσει τα δικαιώματα τα οποία μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας και τα οποία έχουμε υπερψηφίσει στην Επιτροπή το ότι γίνονται ψηφίσματα με μία ψήφο εναντίον ε, είναι γεγονός. Δυστυχώς κανένας από τους πράσινους δεν ήταν παρόν στην ψηφοφορία. Εφόσον λοιπόν έχουμε το δικαίωμα βάσει της ε, συνθήκης της Λισαβόνας και το λέει ξεκάθαρα η συνθήκη, όπως είπε ο Πέτερ Γιάρ, εμείς απλώς ε, χρησιμοποίησαμε τα δικαιώματα, τις αρμοδιότητες που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας. Έχουμε το δικαίωμα της συναπόφασης και αν δεν το χρησιμοποιήσουμε βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας δεν επιτελούμε σωστά το έργο μας. Πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία ε, από την Επιτροπή μας θα δείξει στην Κομισιόν ότι θα πρέπει να συμπεριφέρεται με μεγαλύτερη προσοχή στις πράξεις κατά εξουσιοδότηση έναντι του Κοινοβουλίου. Έχουν ζητήσει το λόγο αρκετοί συνάδελφοι. Θα σας δώσω το λόγο. Σας υπενθυμίζω όμως ότι έχουμε αποχαιρετιστήριο κοκτέιλ. Ε, να είμαστε λίγο σύντομοι ε, για να τελειώνουμε. Μην τσακώνεστε. Ε, ο κύριος Άγνιο. Well, Πρόεδρε, δεν θέλω να εμποδίσω τον κόσμο να πιει, αλλά διαφωνώ με τον Άλμπερτ Ντες. Είπε ότι η Κομισιόν θα επιδείξει μεγαλύτερη φρόνηση τώρα στο εξή για τις κατεξουσιοδότηση πράξη. Εγώ νομίζω ότι δεν θα είναι πιο φρόνιμη, διότι τώρα αρκεί μία κατεξουσιοδότηση πράξη με λίγο αφρό από πάνω και μετά αφήνουν τους ευρωβουλευτές να βγάλουν τον αφρό και μένει αυτό που ήθελαν από την αρχή. Εκπλήσωμε που δεν δεχτήκαμε το 6 γιατί τώρα καταλήξαμε σε κάτι το τελείως ακατάληπτο γιατί τα αρχικά κείμενα είναι τα αγγλικά. Αν στα αγγλικά δεν έχουν νόημα, τότε δεν θα έχουν νόημα και στις μεταφράσεις. Και τουλάχιστον θα μπορώ εγώ να πω ότι προσπάθησα να πείσω τους υπόλοιπους, προσπάθησα να καταψηφίσω και νομίζω ότι είμαι ο μόνος και πρώτος ευρωβουλευτής στην ιστορία του Κοινοβουλίου που θέλησε να καταψηφιστούν οι κατεξουσιοδότης πειράξεις. Ευχαριστώ. στα πλαίσια των ε, κατεξουσιοδότησης πράξεων, για τις κατεξουσιοδότησης πράξεις μάλλον, θα ήθελα να πω ότι δεν πρόκειται για ουσιώδη τμήματα του δικαίου, άρα, άρα λέγω, το θέμα είναι μόνο πώς θα εφαρμοστεί μια πράξη βασικού δικαίου, ενώ οι κατεξουσιοδότης πράξεις δεν μπορούν να τροποποιήσουν το θεμελιώδες αυτό δίκαιο. Αυτό όμως κάναμε εμείς τελικά κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε τον συντελεστή και κατεμένα. ο κανόνας αυτός πρέπει, για τον κανόνα αυτό πρέπει να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί η τροποποίηση αυτή δεν έπρεπε να γίνει με κατεξουσιοδότηση πράξη. Και πρόκειται για προηγούμενο επικίνδυνο διότι οι νομικοί κανόνες που εγκρίνονται από κατεξουσιοδότηση πράξη θα έπρεπε στο μέλλον να μπορούν να τροποποιούνται για να προστατευτεί το καθεστώς συνομοθέτη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. ήταν παράδοξο, παράδοξο από τους συντηρητικούς και ιδιαίτερα από τον Άλμπερντ Ντε στις τελευταίες εβδομάδες όλο αυτό το θέατρο ε, και η συνεργασία με τους αντιπάλους της Ευρώπης, τους ευρωσκεπτικιστές κλπ. Ε, και εν συνεχεία έγινε ένα μπέρδεμα ότι πρέπει να εφαρμόσουμε δημοκρατικές διαδικασίες αλλά αυτή δεν είναι δημοκρατία κλπ. Ή ο Άλμπερντες ο υπεραμείνεται της μεταρρύθμισης και συμφωνεί με την Κομισιόν διότι θα πρέπει, παρόλο που θα μας κατηγορήσουν ότι έχουμε την ευθύνη, ε, να, δεχθούμε τις κατηγορίες. Αλλά το να κατηγορούμε μόνο την Κομισιόν για όλα τα στραβά τα οποία έγιναν, ε, αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Η Κομισιόν ελέγχεται, έτσι δεν είναι. Μετά από ένα χρόνο θα ελεγχθεί όλη η διαδικασία και ο Αλμπερντές και η Μπρίτα πολλές φορές έχουν ψηφίσει μαζί. Ε, είναι παράδοξο συνασπισμός αυτός. Τι να πω, δεν είναι ευρωπαϊκή συμπεριφορά αυτή. Ή δέχεσαι τις ευθύνες σου ως προς την μεταρρύθμιση, αλλά να παίζεις και να κοροϊδεύεις πίσω από τις πλάτες των παραγωγών και των γεωργών είναι απαράδεκτο. Ο πρόεδρος, η Μπρίτα. Λοιπόν, καταρχάς, στην ψηφοφορία υπήρξα συνεπής ως προς τον πρώτο πυλώνα. Δεν άλλαξα τη στάση μου έναντι άλλων πολιτικών ομάδων που τώρα υπερψήφισαν ενώ παλιότερα είχαν καταψηφίσει. Δεύτερον, Μία πτυχή της δημοκρατίας είναι η πλειοψηφία, αλλά υπάρχουν και οι μειοψηφίες οι οποίες πρέπει και αυτές να γίνουν σεβαστές. Τώρα να παρουσιάζουμε, να χρωματίζουμε τις μειοψηφίες ως ε, ε, αντίθετες προς την Ευρώπη είναι απαράδεκτο. Η Ευρώπη δεν είναι δικτατορία. Ε, οι απόψεις της μειοψηφίας και αυτές ανήκουν στο ευρύτερο δημοκρατικό πλαίσιο. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτή η συζήτηση ωφελεί κανέναν, μας βλάπτει. Καλύτερα θα είναι να πούμε ότι είχαμε τη δυνατότητα να εκφράσουμε τις αντιρρήσεις μας ως προς τις πράξεις αυτές και όλοι οι ευρωβουλευτές ψήφισαν κατά συνείδηση. Όχι... Ε, εν συνεχεία ε, να τρέχουμε πίσω από τις ομάδες ε, και τους ε, συναδέλφους μας και να τους κατηγορούμε, αλλά να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Είναι μία γραφειοκρατία την οποία στα πλαίσια της μεταρρύθμισης δεν θα το δεχτώ. Εάν στον πρώτο πυλώνα συμπεριληφθεί το screening, δεν συμφωνώ. Πιστεύω ότι θα έπρεπε στην πρώτο πυλώνα να υπάρξει αυτό το capping, ο περιορισμός του screening και εν συνεχεία να μπει στον δεύτερο πυλώνα. Αλλά το να βγάζουμε εδώ τα άπλητά μας τη φόρα το βρίσκω επιβλαβές. Ευχαριστώ Μπρίτα, ο Τζιμ Νίκολσον και μετά ο Άλμπερτ Ντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω το Ζωζέ για αυτά που είπε, εμείς υποστηρίζουμε αυτή τη θέση ε, ευθύς εξ αρχής υπάρχει μια σοβαρή προειδοποίηση για το Κοινοβούλιο στο μέλλον για τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Εκεί δεν είδε το πρόβλημα σε όλες τις διαπραγματεύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Κάναμε τις διαπραγματεύσεις και η ανησυχία μας ήταν ε, να έχουμε την πολιτική συμφωνία τον περασμένο Ιούνιο. Όταν λάβαμε τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση, σίγουρα δεν αντανακλούσαν αυτό που είχαμε συμφωνήσει τον Ιούνιο και φυσικά εκεί ανησύχησα κι εγώ και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τελείσει κάποια διδάγματα. Είμαστε ε, οι, ε, οι νέοι σε αυτή την υπόθεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ε, έφτασαν στο θέμα των πράξεων κατοξουσιοδότηση εξουσιοδότηση ήταν πάρα πολύ πιο έμπειροι και νομίζω ότι αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, χρειάστηκε να κάνει το ελάχιστο από αυτά που έπρεπε να κάνουν και τα κατάφερε. Και νομίζω ότι αυτό δεν αποκλείει και αυτό που κάνουν τα, μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη σε περιφερειακό επίπεδο για τους γεωργούς. Θα πρέπει να τα εφαρμόσουν όλα αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν ή που θα συμφωνηθούν. Και εκεί διαπιστώνουν ότι αντί να βελτιώσουν την κατάσταση και να έχει λιγότερη γραφειοκρατία, θα υπάρχει περισσότερη γραφειοκρατία και νομίζω θα αρχίσουν να αναρωτιούνται προς τι όλο αυτό και όπως είπε και η Μπρίτα, είναι λίγο αργά τώρα να με ψημιρούμε. Για όσους επιστρέψουν ίσως και στην Επιτροπή Γεωργίας, ε, θα πρέπει να κάνουν κάτι. Ε, υπάρχει μια επιτυχία. Ο Επίτροπος είπε ότι ξεκινούν νέα πράγματα για τη γεωργική παραγωγή και θα ε, επανεξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έγινε μετά από 12 μήνες. Ίσως είναι το καλύτερο που καταφέραμε να επιτύχουμε μακροπρόθεσμα και αυτή η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση θα μας επιτρέψει, ε, μάλλον αντί για μεσοπρόθεσμη ε, αναθεώρηση θα έχουμε νωρίτερα δυνατότητα να εξετάσουμε τα θέματα. Ο Άλμπερτ Ντες, ε, ο Λουίς Καπίλος Σάντον και θα κλείσει η κυρία Γέγκλη. Ευχαριστώ. Ζήτησα το λόγο. Διότι απορρίπτω στεναρά τις παρατηρήσεις του κυρίου Χολστάιν. Εδώ και 30 χρόνια εργάζομαι για την ευρωπαϊκή ιδέα από την ηλικία των 15 ετών υπερμάχομαι της ευρωπαϊκής ιδέας και δεν μπορεί κανένας να με κατηγορήσει ως ενάντιο της ευρωπαϊκής ιδέας. Εγώ πάντοτε εκπροσωπούσα μία συνεπή γραμμή. Αλλά πρέπει να λάβω υπόψη και ε, την ομάδα μου. Και, και εγώ δεν ήθελα το greening στον πρώτο πυλώνα, το ήθελα στον δεύτερο πυλώνα και στο Κοινοβούλιο και στην προηγούμενη Επιτροπή είχαμε λάβει μία απόφαση με μεγάλη πλειοψηφία που έλεγε ότι το Κοινοβούλιο δεν επισημεί νέο σύστημα πληρωμών το οποίο θα οδηγήσει σε νέες ελεγκτικές διαδικασίες και ακριβώς αυτό δημιουργούμε ε, με το greening ε, και γι' αυτό παρέμεινα πιστό στη γραμμή μου σήμερα ε, τρεις, φορ, τρία μέλη ψήφισαν διαφορετικά και θα δείτε τι προβλήματα θα έχουμε στο μέλλον. Είχα συζητήσει με εκπροσώπους της διοίκησης και μου είπαν ότι δεν φταίνε οι, τροπολογίες του ΕΛΚ για περισσότερη γραφειοκρατία για την επιβάρηση της γραφειοκρατίας αλλά οι προτάσεις της Κομισιόν αυτές θα επιβαρύνουν τη γραφειοκρατία θα δείτε λοιπόν τι θα γίνει και η ε, αναθεώρηση της αγροτικής πολιτικής θα ε, είναι αυτή την οποία επιθυμούμε εδώ και 50 χρόνια. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σεβαστές όλες οι απόψεις εδώ μέσα. αλλά αυτό που μετράει είναι οι αποφάσεις και εγώ είμαι περήφανος διότι ως Ευρωβουλευτής βρίσκω ότι το Κοινοβούλιο έπαιξε πολύ θετικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Εκείνοι που έλεγαν ότι αργά ή γρήγορα το Κοινοβούλιο θα έχει δικαιοδοσία συναπόφασης τελικά αποδείχτηκαν σωστή. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την υπεύθυνη στάση που τηρήσαμε σήμερα υπέρ της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, υπέρ των Γεωργών και υπέρ της Ευρώπης. Ευχαριστούμε η κυρία Γέγκλε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ απορώ για τις ε, δηλώσεις ε, των πρασίνων συναδέλφων. Κύριε Ρόσλι, ποτέ φορές ε, στις, στα 15 χρόνια με, με έχει ξεφωνήσει κάποιος ε, ε, ένα υπουργικό στέλεχος όσο στο τηλέφωνο. Με, με, με τρέλανε στις φωνές, ε, τηλεφωνικός δηλαδή στη Βαβαρία, σε έξαλλη κατάσταση. Και παρόλα αυτά, παρόλα αυτά, εγώ είπα ότι δεν υποχωρώ. Έχουμε μία πολιτική ένωση και ε, διάβασα με πολύ προσοχή, ενώ εσείς σίγουρα δεν διαβάσατε, ε, το, την ουσία των τροπολογιών μου. Με πολύ προσοχή μελέτησα τις τροπολογίες μου και είδα ότι από το νομικό πλαίσιο υπάρχει μία διαφορά και αυτή η ε, διαφορά δεν ε, αναφέρεται μόνο στη βασική δήλωση αλλά πάει και πολύ πιο πολύ προχωρεί εις βάθος. Αυτές οι αλλαγές δηλαδή είναι πολύ ευρύτερες. Έχουμε λοιπόν και το δικαίωμα και το καθήκον βάση της Λισαβόνας να εξετάσουμε αυτά πολύ προσεκτικά αυτές τις πράξεις. Μετά από 15 χρόνια, Πρόεδρε, αυτή ήταν η τελευταία μου παρέμβαση. ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την συνεργασία τους αυτά τα 15 χρόνια. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία, ευχαριστώ και τη δική σας Προεδρία ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Επιτροπής τα τελευταία χρόνια. Ε, ευχαριστώ, Ελιζαμπέθ. Ο Ζωζέ θέλει το λόγο. Δύο λόγια. Δεν θέλω να ξαναρχίσω διαμάχες. Ε, δεν επιτίθεμε ε, κατά των γεγονότων και κατά των ε, ατόμων και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές. Για μένα πρόκειται για μια πραγματική πολιτική συζήτηση για τις διάφορες επιλογές που γίνονται. Ο Άλμπερντ Ντές ήταν απόλυτα σαφής και τον ευχαριστώ για την τελευταία του παρέμβαση, διότι μας είπε ότι όλα όσα έκανε προκειμένου να σαμποτάρει την τελευταία πρόταση έγιναν για να επιτεθούμε στο greening ε, στον πρώτο πυλώνα. Όλα λοιπόν εκεί ε, συνοψίζονται. Για μένα είναι σαφή, δεν υπάρχει καμία αμφισημία. Θεωρώ ότι η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε ε, δεν είναι και τόσο συνηθισμένη αν θέλετε, αλλά αυτό είναι ένα πολιτικό παιχνίδι και ε, αλλάζουν τα πράγματα. Δεν έχω πρόβλημα και θα ήθελα να πω, γιατί νομίζω ότι η κυρία ε, Ρέιμερς δεν κατάλαβε αυτά που είπα. Ε, η ομάδα της ήταν συνεπής σε αυτά τα οποία υποστήριζε. Δεν έχω πρόβλημα με την ψηφοφορία. Η ουσία του προβλήματος ε, ε, είναι αυτό το οποίο με απασχολεί. Η οικολογική συνιστόσα, αυτή η πράσινη συνιστόσα και η ρήτρα ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, δυνατότητα ενός χρόνου ε, μετά από τον οποίο θα γίνει αξιολόγηση, σημαίνει ότι όλα όσα ψηφίζαμε σήμερα είναι προσωρινά. Ούτε μακροπρόθεσμα δεν θα μπορούμε να δούμε τις συνέπειες της νέας γεωργικής μας πολιτικής. Και νομίζω ότι εδώ είναι ο μεγάλος κίνδυνος και ελπίζω όλοι όσοι βρίσκονται στην αίθουσα να βρίσκονται και στην επόμενη συνεδρίαση της 7ης Ιουλίου εδώ και να αντιληφθούν ότι ίσως κάναμε κάποιο λάθος και ε, να προσπαθήσουμε μετά τις διακοπές και μετά τις ευρωεκλογέ να ξεκινήσουμε με νέα όθηση. Ήταν χαρά μου να συνεργαστούμε με όλους σας και ελπίζω να είμαστε όλοι εδώ μαζί τον Ιούλιο. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο καθής εξέφρασε την άποψή του. Ήταν ε, συναρπαστικά αυτά τα χρόνια. Νομίζω καταφέραμε να περάσουμε αρκετή νομοθεσία και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ε, διστάμενε απόψεις αρκετές φορές, καταφέραμε να έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα και συμφωνώ με αυτά που είπε ο Λουίς Καπούλες. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για το ρόλο του Κοινοβουλίου, γιατί σίγουρα είχαμε τη δυνατότητα να αποδείξουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει αποτελεσματικό ρόλο. Σίγουρα θα ήθελαν κάποιοι από εμά ε, μια διαφορετική μεταρρύθμιση, αλλά τα καταφέραμε και η μεταρρύθμιση έγινε με συμμετοχή όλων και νομίζω ότι αυτό ήταν προφανές σε όλο το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή μας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και το ξέρουν όλοι. Σας ευχαριστώ. Είναι η τελευταία φορά που μιλώ εδώ ως πρόεδρος. Χάρηκα ιδιαίτερα. Θα τα πούμε τώρα όλα διαζώσεις με ένα ποτηράκι κρασί και για την υποστήριξή σας και για τις διαφορές και φυσικά να ευχηθώ σε όλους ε, στο επαναδείμ. Να δώσω τώρα το λόγο στον Αλμπερτές που έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα πρέπει πριν λήξει η συνεδρίαση θα, ως πρόεδρος του ΕΛΚ και εκ μέρου των συναδέλφους θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, το προεδρείο, τον αντιπρόεδρο, όλους τους συναδέλφους Ευχαριστώ τους πάντες χωρίς να αποκλείω κανέναν για την πενταετή συνεργασία και χαίρομαι που καταφέραμε ε, πολλά, πολλά από κοινού, ε, πολλές αποφάσεις λήφθησαν με ομοφωνία και αποχαιρετώ θερμά και όλους τους συναδέλφους που δεν θα είναι στην επόμενη θητεία, ε, τους συναδέλφους που δεν θα ε, υποβάλουν εκ νέου υποψηφιότητα, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα και ευχαριστώ και εσάς Πρόεδρε για τη μακροχρόνια συνεργασία σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Άλμπερτ. Επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας προβλέπεται για τις 7 Ιουλίου για όλους όσοι θα είναι ακόμα εδώ ε, σας ευχαριστώ, καλή τύχη, καλή προεκλογική εξαιρετία και θα τα πούμε εδώ απ' έξω για ένα ποτηράκι.